Γιατί βέβαια τα ίδια προβλήματα έχουμε στη γειτονιά μα και στα ανατολικά μα, όχι μόνο προ το νότο. Και θα πρέπει οι πολιτικέ που ακολουθούμε να είναι υπεύθυνε και να μην βασίζονται μόνο στα συναισθήματά μα, παρόλο που μπορεί να συγκινούμαστε πολλέ φορέ σαν άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Μια και έχουμε μείνει πολύ πίσω, ε, θα επιτρέψω την τελευταία μπλε κάρτα για την συζήτηση αυτή, γιατί πραγματικά δεν έχουμε χρόνο για να παρατείνουμε περαιτέρω τη συζήτησή μας. Ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, ε, Ρασίτα Μπιελάμι από τη Βουλή του Μαρόκου βρίσκεται στον εξώστη και παρακολουθεί τις εργασίες μαζί με αντιπροσωπεία. Τους καλωσορίζουμε και ελπίζουμε να είναι ενδιαφέρουσα και καρποφόρη η επίσκεψή σας. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστεί και στα γαλλικά ο πρόεδρος.